Καλημέρα. Κυρίσω την ε, έναρξη της συνεδρίασης. Και πριν προχωρήσουμε στις ε, διάφορες συζητήσεις που προβλέπονται στην ημερήσια διάταξη, έχω να ανακοινώσω τα αποτελέσματα της δεύτερης ε, περίοδου ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα αυτά λοιπόν, της Τετάρτης δηλαδή, έχουν ως εξής. Πρώτον, είχαμε ε, κάποιες ενιαίες ψηφοφορίες. Η πρώτη για το Κάπο Βέρντε, που εγκρίθηκε. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα συμβουλευτείτε και στην οθόνη. Εγκρίθηκε λοιπόν το Κάπο Βέρντε. Στη συνέχεια είχαμε και άλλο ψήφισμα για το Κάπο Βέρντε που εγκρίθηκε. Στη συνέχεια είχαμε δύο πρωτοβουλίες για την Γουινέα Μπισάου που εγκρίθηκαν και οι δύο. Στη συνέχεια είχαμε πρωτοκόλλο για το Σάντο Τομέ, εγκρίθηκε και αυτό. Και μετά πρωτοβουλία για την ε, Ελβετία που εγκρίθηκε. Είχαμε επίσης μία πρωτοβουλία για την κεφαλοπάθεια που εγκρίθηκε και αυτή. και άλλη ενιαία ψηφοφορία για το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης, αντιμετώπισης της παγκοσμιοποίησης. Ε, εγκρίθηκε όπως επίσης και το Ταμείο Αλληλεγγύης. Επόμενη πρωτοβουλία που εγκρίθηκε είναι ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2020. Πρωτοβουλία για τη Μολδαβία επίσης εγκρίθηκε, πρωτόκολλο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας επίσης εγκρίθηκε. Ε, στη συνέχεια είχαμε πρωτοβουλία για το Μαρόκο που εγκρίθηκε. Πρωτοβουλία για την Ιορδανία που εγκρίθηκε επίσης. πρωτοβουλία για την Κίνα που εγκρίθηκε. Επίσης πρωτοβουλία για τη Γεωργία εγκρίθηκε. Και τέλος, πρωτοβουλία για την ε, συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Εγκρίθηκε επίσης. Τώρα, έχω να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα ε, τα σχετικά με τις τροπολογίες. Τροπολογίες της προτάσεις ψηφίσματος. Ε, διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. 18. Τα βλέπετε και στις οθόνες. Η τροπολογία 18 λοιπόν απορρίφθηκε. Τροπολογία αριθμός 1 απορρίφθηκε. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε και στην ε, οθόνη σας. Τροπολογία αριθμός 2 απορρίφθηκε. Τροπολογία 3 απορρίφθηκε. Τροπολογία 11. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 19. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 20. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 4. Απορρίφθηκε. Τροπολογία αριθμός 5. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 6. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 7. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 21. Απορρίφθηκε. Στη συνέχεια έχουμε Παράγραφος 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε. Τροπολογία αριθμός 8. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 22. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 23. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 12. Απορρίφθηκε. 13. Για την αιτιολογική σκέψη α. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 14. Απορρίφθηκε. Αιτιολογική σκέψη Β. Πρώτο τμήμα. Εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη Β. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 15. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 16. Απορρίφθηκε επίσης. Τροπολογία 17 στην αιτιολογική σκέψη Δ, επίσης απορρίφθηκε. Τώρα θα σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα όσον αφορά τα ψηφίσματα για τις ειδικές ε, επιτροπές. Πρώτα απ' όλα για την Ειδική Επιτροπή για την ανάμειξη στα εξωτερικά. Πρώτη τροπολογία απορρίφθηκε. 7. Απορρίπτεται. 8. Απορρίπτεται. 9. Απορρίπτεται. 2. Απορρίφθηκε. 10. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 3. Απορρίφθηκε. 11. Απορρίφθηκε. 12. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 4. Απορρίφθηκε. 13. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 5 δέλτα. Απορρίφθηκε. 14. Απορρίφθηκε. 16. Απορρίφθηκε. 6. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 6 απορρίφθηκε. Έξι, ένα, αλφα, απορρίφθηκε. Διορθώνει ο πρόεδρος. Έχω ήδη περάσει σε άλλη πρόταση για την ειδική πρόταση όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εδώ υπάρχει πάλι μια τροπολογία αριθμός 6 που απορρίφθηκε. Τροπολογία 7. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9 Δέλτα. Απορρίφθηκε. 13. Απορρίφθηκε. 10 Δέλτα. Απορρίφθηκε. 14. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 15. Απορρίφθηκε. Τροπολογία αριθμός 1. Απορρίφθηκε. 2. Απορρίφθηκε. 11. Απορρίφθηκε. 3. Απορρίφθηκε. 4. Απορρίφθηκε. 12. Απορρίφθηκε. 5. Απορρίφθηκε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για δημιουργία ειδικής επιτροπής όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη. Και τώρα περνάμε στις ε, διορθώσεις όσον αφορά το COVID-19. Τροπολογία 5. Εγκρίθηκε. Τροπολογίες 1 και 4 απορρίφθηκαν. Τροπολογία 2. Απορρίφθηκε. 3. Απορρίφθηκε. Τώρα, εδώ ολοκληρώνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου ψηφοφοριών που διεξήχθη εχθές. Τώρα λοιπόν που σας ανακοίνωσα τα αποτελέσματα μπορούμε να περάσουμε και στις συζητήσεις που προβλέπονται για σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Όπως γνωρίζετε θα ξεκινήσουμε με μια κοινή συζήτηση Έχουμε δηλώσει του Αντιπροέδρου τη Επιτροπή και είπα του εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Τον οποίο και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του εδώ. Έχουμε δηλώσεις λοιπόν για τα εξή θέματα. Επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στην εξωτερική πολιτική. Νομοθεσία της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας περί εθνικής ασφάλειας για το Χονγκ Κόγκ και η ανάγκη να υπερασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κόγκ και αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της δυτικής όχθης από το Ισραήλ. Θέλω να επενθυμίσω στους ευρωβουλευτές ότι σε αυτή την κοινή συζήτηση δεν θα έχουμε αυθόρμητες παρεμβάσεις και ούτε μπλε κάρτα. Ούτε κατσδιά, ούτε μπλε κάρτα δηλαδή. Οπότε δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπατε εκπρόσωπο τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, τον κύριο Μπορέλ και τον ευχαριστώ και πάλι που βρίσκεται εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Μπορέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές. Τρία είναι τα ζητήματα και θα αναφερθώ αμέσως σε αυτά. Πρώτα απ' όλα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση του κορονοϊού. Είναι σαφές ότι μια παγκόσμια πανδημία όπως αυτή χρειάζεται και παγκόσμιες λύσεις και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στο επίκεντρο αυτών των απαντήσεων. Τον Απρίλιο λοιπόν ξεκίνησε μια προσπάθεια για να βοηθήσουμε τις χώρες εταίρους που αντιμετωπίζουν την πανδημία. Έχω ήδη παρουσιάσει τα σχετικά στοιχεία στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Στις 6 Ιουνίου συζητήσαμε στο ε, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για τον τομέα της ανάπτυξης που μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα ε, και κινητοποίησαμε 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες χώρες ε, της Αφρικής ε, στη γειτονία μας. Ε, δεν είναι βέβαια καινούριο χρήμα αυτό. Είναι χρήματα τα οποία έχουν ήδη διατεθεί και τα οποία ε, επαναδιαθέτουμε. Ήταν όμως πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα της πανδημίας. Τώρα, τα προγράμματα για τους πρόσφυγες, τα οποία επεκτείνονται, κρίσιμο και αυτό. Εμείς καλωσορίζουμε τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε τον, που θα, θα εγκρίνει τον Ιούλιο μάλλον ε, το περαιτέρω αυτά κονδύλια 400 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη των, ε, των προγραμμάτων για τους πρόσφυγες. Επίσης για την εξωτερική δράση και σχετικές πολιτικές ε, έχουμε ένα top-up για το, στα πλαίσια του εργαλείου Next Generation της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μέρος αυτού του ποσού θα πάει στην ανθρωπιστική βοήθεια ένα άλλο σε, μια υψηλότερη οροφή για την εγγύηση της εξωτερικής δράσης στα πλαίσια ε, του οργάνου για την ε, ανάπτυξη της γειτονίας και της στρατηγικής συνεργασίας προβλέπεται, και περαιτέρω 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, έτσι ώστε να παράσχουμε εγγυήσεις έως 130 δισεκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης ε, καθώς και περαιτέρω μικροοικονομική ενίσχυση ε, για τις τρίτες χώρες. Αυτό θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε ε, τη βιώσιμη και την πράσινη ε, δέσμοι επενδύσεων ε, στις χώρες αυτές. Ελπίζω να μας υποστηρίξετε για να έχουμε ένα φιλόδοξο επίπεδο πόρων στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, να πω βέβαια ότι είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, έτσι, διότι αυτή η κρίση θα έχει βιβλικές επιπτώσεις. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική, παραδείγματος χάρη, όπου τα πράγματα χειροτερεύουν στην Αφρική ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο θα ανέμενε κανείς αλλά οι υγειονομικές αλλά οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι σημαντικές ούτως ή άλλως και δυστυχώς ε, φοβάμαι ότι θα κρατήσουν και μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο ζήτημα ε, στη σημερινή συζήτηση έχει να κάνει με την Κίνα και την ε, σχετική νομοθεσία για το Χονγκ Κόνγκ. Θέλω να πλαισιώσω την απάντησή μου πάνω στο εξή γεγονός. Το COVID έχει επιταχύνει τις υπάρχουσες τάσει. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθημερινά αυξανόμενη ένταση. Θέλω να επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλάκι στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τον δικό της τρόπο για, για να ισορροπήσει στη σχέσεις της και με τους δύο αυτούς παράγοντες. Ο Γάλλος υπουργό εξωτερικών έλεγε λίγο πολύ χθε ε, τα ίδια πράγματα στον γαλλικό τύπο ε, και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο, μια άποψη την οποία μάλλον συμμεριζόμαστε και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ίσες αποστάσεις. Η διατλαντική συμμαχία, η διατλαντική υπερική σχέση είναι, είναι η πιο σημαντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βεβαίως και έχουμε αποκλήσει με την υπάρχουσα κυβέρνηση ε, στο, ΗΠΑ. Αυτό είναι προφανές για μια σειρά αποζητήματα σε ό,τι αφορά τη θέση τους για την πολυμερή προσέγγιση, σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη το παγκόσμιο, ε, το διεθνές μάλλον ποινικό δικαστήριο, αλλά όποτε είναι δυνατόν θέλουμε να έχουμε θετικέ σχέσει. Η σχέση μα τώρα με την Κίνα δεν μπαίνουν, ε, δεν μπορούν να περιγραφούν απλά. Δεν είναι μια απλή σχέση. Είναι μια περίπλοκη σχέση. Δεν μπορούμε να απλουστεύουμε, υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα. Χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται αμοιβαιότητα, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Η Κίνα είναι ένας εταίρος απαραίτητος, είτε μας αρέσει είτε όχι, για να επιλύσουμε κάποια παγκόσμια ζητήματα, όπως η πανδημία, παραδείγματος χάρη, η κλιματική αλλαγή. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορούμε να επιλύσουμε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής χωρίς σημαντική δέσμευση από τους Κινέζους. Ταυτόχρονα, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν ένα κρίσιμο, ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στις σχέσεις μας. Έθεσα το θέμα των, της κατάστασης στο Χονγκ Κόνγκ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε μια μακρά συζήτηση, πάνω από τρεις ώρες, πρόσωπο με πρόσωπο. Ε, ήταν πιστεύω χρήσιμη και ειλικρινής αυτή η συζήτηση, ανοιχτή για όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιπλοκή σχέση μας και βεβαίως ε, αυτή η νομοθεσία περί ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ δεν συνάδει με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κίνα ιδιαίτερα ε, στα πλαίσια της κοινή δήλωσης Κίνας Ηνωμένου Βασιλείου ε, που περιλαμβάνεται στην νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ. Η αυτονομία του Χονγκ Κονγκ και τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χονγκ Κονγκ μας αφορούν και εμά άμεσα. Είναι θέμα αξιών, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα σεβασμού διεθνών δεσμεύσεων δεν μπορούμε να υπονομεύουμε έτσι ε, την αρχή του μία χώρα, δύο συστήματα και την αυτονομία του Χονγκ Κόνγκ. Ε, όπως γνωρίζετε το είπα σαφώς αυτό στη δήλωσή μου στο όνομα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 και 29 Μαΐου και βεβαίως ομόφωνα αποφασίστηκε αυτό κάτι που συμβαίνει όλο και πιο σπάνια στις συζητήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έδωσα το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όταν είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ εκεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ίδια μέρα που πάρθηκε αυτή η απόφαση. Και είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως στη συνέχεια κατά τη κατά τις να αναφερθώ στις διάφορα, διάφορα μέτρα που, έχω, που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα αυτό. Το τρίτο ζήτημα τώρα. Η ενδεχόμενη προσάρτηση της δυτικής όχθης του Ιορδάνη από τους Ισραηλινούς ε, από το Ισραήλ μέρος ε, των κατεχομένων Παλαιστινιακών εδαφών. Εδώ η θέση μας είναι σαφής. Παρότι για άλλη μια φορά είναι δύσκολο να βρεθεί ομοφωνία. Υπάρχει όμως ε, μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία κρατών μελών που εξακολουθούν να υποστηρίζουν ε, μια λύση δύο κρατών μετά από διαπραγμάτευση με βάση διεθνείς παραμέτρους και θεωρούν βεβαίως ότι η προσάρτηση, οποιαδήποτε προσάρτηση ε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Έτσι λοιπόν ζητούμε από το Ισραήλ να μην προβεί σε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την προσάρτηση οποιοδήποτε εδάφους Παλαιστινιακού. Είχα την ευκαιρία να εκφράσω την άποψη αυτή στη τηλεφωνική συνομιλία με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών και Άμυνα του Ισραήλ. Του νέου Υπουργού Εξωτερικών και Άμυνα του Ισραήλ. Ε, πρόκειται για σοβαρή παραβίωση, παραβίαση του διεθνού δικαίου εδώ. Τον Μάρτιο στη Γενέβη 27 κράτη-μέλη συμφώνησαν επ' αυτού. Στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών δεν φτάσαμε σε ομοφωνία δυστυχώς επί του ίδιου ζητήματος, αλλά όπως είπα μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία κρατών μελών εξακολουθεί να υποστηρίζει αυτήν την αρχή. Ε, δεύτερον, αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη ζημιά στην προοπτική μιας λύσης με, που θα βασίζεται στα δύο κράτη θα επηρεάσει την περιφερειακή σταθερότητα, την σχέση μας με το Ισραήλ, τη σχέση του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες και βεβαίως και την ίδια την ασφάλεια του Ισραήλ που είναι κάτι το οποίο είναι μη διαπραγματεύσιμο για μας. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Τέλος, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσάρτηση ε, θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις ε, και ε, στη συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ δεν θέλω να ξεπεράσω το χρόνο που μου αναλογεί. Ε, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στον ενδεχόμενο αντίκτυπο μια προσάρτηση. Πάντω η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τι ευθύνε τη ε, με βάση το διεθνέ δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και όπω αποφασίστηκε στα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων μέσα Μαΐου, με το Ισραήλ προσπαθούμε να αποφύγουμε να συμβεί αυτό, να γίνει αυτό το βήμα πριν είναι πολύ αργά. Χρησιμοποιούμε κάθε διπλωματικό μέσο για να, για να ασκήσουμε πίεση ώστε να μην συμβεί αυτό. Ε, επικοδομητικές συζητήσεις βεβαίως θέλουμε να έχουμε με τον ε, κύριο Γκάντ, τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Σκενάζη, τον Υπουργό Εξωτερικών και εκεί ε, τους είπα ακριβώ το που σας είπα εδώ τώρα πόσο σοβαρό θα ήταν ένα τέτοιο βήμα. Είμαι βεβαίω και σε στενή επαφή με τι παλαιστινιακέ αρχέ. Ε, πολλοί Υπουργοί Εξωτερικών έστειλαν το ίδιο μήνυμα. Είχαμε μια σημαντική συζήτηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάικλ Πομπέο, αυτήν την εβδομάδα. Και ένα μεγάλο μέρο ε, τη συζήτηση με τον κύριο Πομπέο αφορούσε το Παλαιστινιακό. Τι επόμενε εβδομάδε, του επόμενου μήνε θα συνεχίσουμε να συζητούμε με τι εμπλεκόμενε πλευρέ. Η διεθνή κοινότητα ε, θέλει να υποστηρίξει μία διαπραγμάτευση για μια λύση δύο κρατών με βάση διεθνείς παραμέτρους με ίσα δικαιώματα για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε ε, λίγο περισσότερο χρόνο. Κάπου εδώ θα σταματήσω. Νομίζω ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου. Είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω στα πολλά ερωτήματα που θα έχετε να μου θέσετε. Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, δηλώσεις σας, ε, για αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στους ευρωβουλευτές ε, σύμφωνα με τον κανονισμό να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε τον χρόνο και δεύτερον, να σας παρακαλέσω να παραμείνουμε εντό των θεμάτων που έχουμε. Ξεκινάμε τον κύριο David Μακάλιστερ από το ΕΛΚ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι πεπισμένος για το ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την πρόθεση των συμφερόντων μας σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Οπότε καλωσορίζω την ε, σημερινή συζήτηση για τις συνέπειες της πανδημίας του COVID-19. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η πανδημία δεν θα έχει μόνο ιατρικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές ε, με τρομερές διαστάσεις, αλλά όπως είπε και ο κ. ο αντιπρόεδρος, θα αλλάξει και την γεωπολιτική. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Βλέπουμε μια επιδείνωση της κατάστασης δημοκρατίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυξανόμενες εκστρατείες παραπληροφόρησης και τάσεις απομονωτισμού αντί για συνεργασίες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πως οι νέες αυτές απειλές ε, απαιτούν έντονα και συντονισμένα μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν τους επόμενους μήνες οι επιτροπές που ασχολούνται με τα εξωτερικά να ασχοληθούν με την παγκόσμια αντίδραση. Με την σημερινή συζήτηση αλλά και τις εκθέσεις που απασχολούν τις επιτροπές μας ελπίζω να μπορέσουμε να τονίσουμε την σημασία της εξωτερικής διάστασης και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης με τους ε, εταίρους μας ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, David. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον τον Ινοπίκουλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είπατε πρόσωπε. Οι επιπτώσεις του covid 19 στα διεθνή είναι πολλές από το διεθνές ε, εμπόριο μέχρι την πολυμερή τάξη. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας για να ηγηθούμε τις παγκόσμιες μάχες κατά της πανδημίας με βάση τις δικές μας αξίες και αρχές. Οι προτεραιότητες μας θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τις ευπαθείς κοινότητες, να προωθήσουμε την προσπάθεια για ένα εμβόλιο, την κατάβαση του πυρός και να παραμείνουν ανοιχτές για όλους οι οδοί του παγκοσμίου εμπορίου. Βεβαίως δεν πρέπει να αμελούμε και τα συμφέροντά μας. Αναμένουμε λοιπόν τη νέα ανακοίνωση και θέλουμε να ενισχύσει την ανθεκτικότητά μας. Τέλος, στο πνεύμα της στενής συνεργασίας ε, με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η G20 θα πρέπει να βοηθήσουμε τους διεθνείς εταίρους μας ε, και να οδηγήσουμε ακριβώς ε, την ανάκαμψη μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα τον λόγο για ε, δύο λεπτά στον κύριο Σμάνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή της ε, θητείας η Κομισιόν ανακοίνωσε πως έχει γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Η Ευρώπη θα γινόταν παγκόσμιος παίκτη. Ο κορονοϊός βεβαίως δοκιμάζει αυτές τις φιλοδοξίες. Τους τελευταίους μήνες αναγκαστήκαμε να, δούμε, να περιοριστούμε στα σπίτια μας ε, από τον ιό. Παρόλα αυτά, ο ιός πλέον είναι μια παγκόσμια πρόκληση που φτάνει σε κάθε χώρα του κόσμου. Αυτό μας δείχνει πόσο αλληλένδετοι είμαστε και πόσο αλληλοεξαρτώμενοι είμαστε. Όμως, φαίνεται περίεργο και καθαρά ιδεαλιστικό να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να ενωθούμε παγκοσμίω. Δυστυχώ βλέπουμε χώρε να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή για να διχάσουν την Ευρώπη και να δράσουν κατά των συμφερόντων μα. Για την λεγόμενη κορονοδιπλωματία τη εκστρατεία παραπληροφόρηση, αλλά και την αύξηση της έντασης στην Λιβύη και στην Κίνα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος συνεχίζει να γυρνάει και γρήγορα έχει φτάσει η στιγμή η Ευρώπη να κινηθεί πιο αποφασιστικά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ε, με μια ξεκάθαρη ενωμένη φωνή. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή η Κομισιόν να ανταποκριθεί στις γεωπολιτικές φιλοδοξίες της. Με έναν ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια κοινότητα, με τα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους και όλον τον κόσμο, όπως επίσης και με το εμβόλιο και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους φιλελεύθερους δημοκρατικούς ε, συμμάχους μας στον κόσμο. Ελήψη παγκόσμια ηγεσία από τη ΣΥΠΑ, αυτό τον ρόλο πρέπει να τον παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ε, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει την διαφορά και μπορεί να το κάνει εάν κινηθεί με μια ανανεωμένη αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο Μαρκό Ντρέωστο για ένα λεπτό. Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε Μπορέλ, η κρίση αυτή, όπως είναι σαφές, έχει δημιουργήσει γεωπολιτικές ανισορροπίες. Και βεβαίως ε, η Κίνα δεν συμπεριφέρθηκε ως αξιόπιστος εταίρος κατά τη διάρκεια της κρίσης και δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε την σιωπή. Εμείς επαναλαμβάνουμε δυνατά, όπως το έχει πει και ο πρόεδρός μας, ο Ματέο Σαλβίνη, για μια διεθνή έρευνα για τις αιτίες του ιού. Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας θα πρέπει να δεχθεί αυτή την έρευνα και βεβαίως εσείς ως ύπατος εκπρόσωπος έχετε μεγαλύτερο λόγο από ότι εγώ. Βεβαίως ε, Δυστυχώ η κυβέρνηση των ε, Πέντε Αστέρων και ο Υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι Δημάιο δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα για να σταθούν απέναντι στην Κίνα. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η διαφορά μεταξύ του ελεύθερου και του μη ελεύθερου. Αυτού ο οποίος επιλέγει την ελευθερία και αυτού ο οποίος θεωρεί ότι το ΚΚ της Κίνας είναι ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπουτικόφερ τώρα. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η βασική κρίση η οποία έχει αρπάξει την, ε, τον κόσμο ολόκληρο είναι Βέβαια, ο COVID-19 αλλά είναι και δύο νέα στοιχεία. Είναι η πρώτη διεθνής κρίση που έχουμε εδώ και δεκαετίες όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε αποσύρονται από οποιοδήποτε ηγετικό διεθνή ρόλο ενώ η Κίνα βρίσκεται στο κέντρο της κρίσης αυτής περισσότερο από ποτέ. Και τόσο το καλύτερο. Η κατάσταση αυτή δείχνει ποια είναι η κατάσταση στις διεθνείς σχέσεις. Από την ε, μια βλέπουμε τον αγώνα μεταξύ δύο υπερδυνάμεων και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι διεθνείς θεσμοί είναι αδύναμοι, οι πολυμερείς και είναι αδύναμοι μπροστά στην κρίση και οι τάσεις αυτές επιταχύνονται. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταθεί στο ύψο τη και να φροντίσει να τηρηθούν οι διεθνεί υποχρεώσει. Αποτύχαμε όταν επιβάλαμε απαγορεύσεις στις εισαγωγές-εξαγωγές ή όσον αφορά την έρευνα για τα εμβόλια ή για την συμβολή στον ΠΟΗ που ήθελε μεγαλύτερη βοήθεια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για τις αξίες μας, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας. Τώρα έχω μια παρατήρηση για το Χονγκ Κόνγκ. Ε, χαίρομαι για την δήλωση του G7. Στο ψήφισμά μας λέμε ότι θέλουμε η Κίνα να καταλάβει ότι πρέπει να τηρεί τις διεθνείς της Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Και αυτό είναι που πρέπει να τονίσουμε και την Δευτέρα στη διάσκεψη. Ευχαριστούμε πολύ. Βίτερ Μπατζικόφσκι τώρα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωποι. Πριν από 20 χρόνια, Υπουργός Εξωτερικών ε, μαζί με τον ε, ομολογό του των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν στην Πολωνία. Και σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Και τότε είχε προσκληθεί ο επικεφαλής της Πολωνίας τότε στο Λευκό Οίκο. Τώρα σίγουρα θα συζητηθούν ε, πράγματα γιατί επαναλαμβάνεται η επαφή αυτή μεταξύ άλλων και διατλαντικές σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι υπέρ μια τέτοια συνεργασία. Δεν πρέπει να διχαστούμε, ούτε πρέπει να απομακρυνθούμε από τι ΗΠΑ. Δεν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην Κίνα και τι ΗΠΑ μαζί, να καταπολεμήσουμε τον ιό, την κρίση και να φροντίσουμε για ασφάλεια. Και γι' αυτό κάνω έκκληση σε εσά, κύριε Μπορέλ, και στι υπηρεσίε σα και στις ε, υπηρεσίες εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεισφέρεται στις προσπάθειες που κάνει η Πολωνική Προεδρία ώστε να διασφαλίσει ότι θα ενισχυθούν οι διατλαντικέ σχέσεις και δεν θα πληγούν. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντεμιρέλ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για την κορώνα εδώ και μίες και η πανδημία αυτή μας δείχνει ξεκάθαρα τα λάθη που υπάρχουν στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Εδώ και δεκαετίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τις ιδιωτικοποίησεις. Ε, μόνο από το 2011 έως 2018 ε, είχαμε 63 εκκλήσεις προς τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίησεις της υγείας και από την άλλη στο πλαίσιο της εδωμένης συνεργασίας να αυξήσουν στρατιωτικές δαπάνες. Κύριε Μπορέλ, εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Χάνουν την δουλειά τους ή το εισόδημά τους. Και τώρα ειδικά θέλετε για πρώτη φορά να δοθεί από τον κοινωνικό προϋπολογισμό ένα ποσό 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για έρευνα όπλων, παρά το, άρθρο, παρά το, το άρθρο 41.2 το απαγορεύει ρητά. Γιατί δεν θέλετε να αντιληφθείτε ότι δεν τρώγονται οι βόμβες και τα τεθωρακισμένα. Λέτε ότι ε, η αφελής Ευρώπη πέρασε εγώ λέω ότι είναι αφελές να νομίζουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε μια κούρσα εξοπλισμών. Και δεν είναι αυτός ο τρόπος για να έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο. Κομίν ή Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί το παράδειγμα, πρέπει να καταπολεμήσει την πανδημία, αλλά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει σαν άλοθη για να καταπιέσει το κράτο δικαίου. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο η εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κυριαρχείται από τι βασικέ αρχέ, δηλαδή την στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι δημοκρατικέ αρχέ. Είναι αναγκαίο οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στον κόσμο να μπορούν να αξιοπιστεί να υποστηρίζουν τις αρχές αυτές. Αυτή τη βδομάδα διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια έγγραφα του 80 της ΙΑ που λέει ότι η, κυβέρνηση της Ισπανίας επί έφτιαξε μια ομάδα μισθοφόρων για να καταπολεμήσει εκτός νόμου την τρομοκρατία. Την τρομοκρατία του κράτους όμως εμείς προσπαθούμε ξανά και ξανά να μιλήσουμε και πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και βρίσκονται στη φυλακή. Διακόπτεται το μικρόφωνο του ομιλητή. Ο πρόεδρος το διακόπτει και του λέει «Σας παρακαλώ, οι ομιλητές πρέπει να μιλάνε για τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη, όχι εκτός ημερήσιας διάταξης». Οπότε σας παρακαλώ ολοκληρώστε. Με κάθε σεβασμό, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την πολιτική και την ηθική πτυχή, κύριε είπατε εκπρόσωπε, εσεί δικαιολογείτε αυτήν την τρομοκρατία του κράτου. Η απάντησή σα ε, θα δείξει κατά πόσο νομιμοποιήσετε να είσαστε εκπρόσωπό μα, αλλά κατά πόσο έχει και εξοπιστεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στη διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τους συναδέρφους μην ξεχνάτε ότι έχουμε τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη που συζητάμε τώρα. Παρεμβάσεις για θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιβαρύνουν ε, περισσότερο την ημερήσια διάταξη και είναι εκτός. Δεν προβλέπεται. Οπότε να τηρείτε την ημερήσια διάταξη. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι οικονομικές συνέπειες της ε, κρίσης ε, οδηγούν σε πολιτική αποσταθεροποίηση κρατών και ολόκληρων περιοχών που ούτως ή άλλως έχουν συγκρούσεις. Κάποιοι ε, παίκτες προσπαθούν να προωθήσουν την ατζέντα τους τη στιγμή που η προσοχή μας είναι στραμμένη αλλού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Κίνα την συμφωνία της με το Ηνωμένο Βασίλειο για το Χονγκ και πρόκειται για μια διεθνή υποχρέωση. Δεν είναι ένα έγγραφο που ανήκει στο ιστορικό παρελθόν. Επίση είναι καλό οι Ευρωπαίοι να ταξιδεύουν στο Ισραήλ ή να κάνουν τηλεδιάσκεψη, ειδικά για να ξεκαθαρίσουν στον αρχηγό τη Κυβερνήσεω εκεί πέρα πώς οι προσαρτήσεις ενάντια στο διεθνέ δίκαιο μπορούν να έχουν πάρα πολλέ ε, συνέπειε τι οποίε ε, δεν μπορεί κανεί να προβλέψει σε κράτη όπως η Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ε, ειδικά προς αυτούς που θέλουν να εδραιώσουν τα αρχικά συμφέροντά τους πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εδώ είναι το λόγο στον κύριο Ούντο Μπούλμαν για ένα λεπτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Μπορέλ, και χωρίς τον κορονοϊό, η φετινή χρονιά θα ήταν ε, μια χρονιά από τις χειρότερες εδώ και δεκαετίες. Πριν από λίγα χρόνια 80 εκατομμύρια άνθρωπα, άνθρωποι αντιμετώπιζαν κίνδυνο επιβίωσης. Ε, φέτος ο αριθμός αυτός θα έφτανε τα 120-130 εκατομμύρια άνθρωπους. Η διαφορά οφείλεται στις ε, καταστροφές του περιβάλλοντος και στις στρατιωτικές συγκρούσεις. Τώρα όμως με τον κορονοϊό θα διπλασιαστεί ο αριθμός αυτός. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν να μην έχουν να φάνε. Πρέπει να κινητοποιηθούν γρήγορα κονδύλια και καλά κάνατε, αλλά έχετε έναν αριθμό του ύψους των προσπαθειών που θα απαιτηθεί για να αποφευθούν οι μαζικοί θάνατοι και μπορείτε να μας πείτε κάτι για την πολιτική κυρώσεων κατά του Ιράν, της Βενεζουέλας. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής, αλλά οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να καταπολεμηθεί και εκεί πέρα η πανδημία και η πείνα, ανεξαρτήτως του τι κάνουν οι άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Ούντο. Χάνα Νόημον για μισή λεπτό. Κύριε Μπορέλα, αγαπητοί συνάδελφοι, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην πανδημία COVID σαν να είναι μια κρίση υγείας. Όμως, συγχρόνως, υπάρχει και η κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία ελοχεύει και αυτό επιδεινώνει την υγειονομική κρίση. δεν σταματάει ο ιός μόνο αν περιορίζουμε τους δημοσιογράφους για παράδειγμα αν χρησιμοποιούν σαν άλοθη το COVID διάφορες κυβερνήσεις για να οδηγούνται σε καταστολή αυτό δεν περιορίζει τον ιό αλλά οδηγεί σε θανάτους πρέπει κάθε περιορισμός να είναι αναλογικός. Θα πρέπει να συνδέεται απευθείας με την υγειονομική κρίση και θα πρέπει οι χώρες να μπορούν να συζητήσουν για αυτά και ο κόσμος, ενώ δεν γίνεται αυτό πάντα. Για να καταπολεμηθεί λοιπόν η κρίση COVID-19 συνολικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την υγειονομική κρίση αλλά και την κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να παρακολουθούμε τη διάδοση της ασθένειας αλλά και της παραβιάσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να ερευνήσουμε και τους θανάτους και τις παραβιάσεις. Να προστατεύσουμε τους γιατρούς μας και αυτούς που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Μπορέλ, η Ευρώπη πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς μιλήσατε έντονα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και οι δράσεις μας να ακολουθήσουν, κοιτώντα και στρεφόμενοι προς τον σημερινό κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σικόρκη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον προηγούμενο μιλή, τον κύριο Βατσακόφσκι, ο οποίος μίλησε ιδιαίτερα θετικά σε ό,τι αφορά ε, την κοινότητα της δημοκρατίας. Ε, πρόκειται για το κίνημα του κύριου Γκέρεμεκ, το οποίο συνέχισα και εγώ αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι η πολωνική κυβέρνηση θα σταματήσει να παραβιάζει το κράτος δικαίου και θα ξαναγίνει παράδειγμα δημοκρατίας, ε, ένα παράδειγμα προς μίμηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το COVID-19, ελπίζω να ιεραρχήσουμε κάπως καλύτερα τις ανάγκες μας ε, και στα πλαίσια της διαχείρισης της κρίσης αυτής γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δίνουν την ελπίδα ότι η διαχείριση θα είναι σωστή και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει ενωμένη, όμως ε, η τεχνητή πολιτική των χαμηλών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών. Πολλές ευκαιρίες λοιπόν, αλλά και πολύ κίνδυνοι και ελπίζω αυτό να το έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κάθλιν Βαμπρέμπτη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, ναι εδώ είμαι. Ε, όπως είπατε και εσείς, ο αντίκτυπος της κρίσης του COVID-19 στη διεθνή σκηνή δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά θα είναι τεράστιος και αυτό το γνωρίζουμε. Παίρνω το παράδειγμα της Κίνας, διότι προφανώς είναι μπροστά μας αυτό το παράδειγμα και πριν την πανδημία είχαμε τεράστια προβλήματα στις σχέσεις μας με την Κίνα. Ανθρώπινα δικαιώματα, εμπορικές σχέσεις, το γεγονός ότι πρόκειται για μια κρατική οικονομία ε, και τα λοιπά. Μετά όμως το COVID-19 αυτά τα, τα προβλήματα ε, εντάθηκαν. Μας βομβάρδισαν με fake news, με ψευδείς ειδήσει. Ε, δεν μας έδωσαν τα στοιχεία που πρέπει να μας δώσουν σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και βεβαίως εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από την Κίνα, ιδιαίτερα για το προστατευτικό υλικό στα, πλαίσια της κρίσης αυτής. Να είστε, είμαστε σαφείς λοιπόν κύριε Μπορέλ, ε, η εμπορική πολιτική είναι το πιο σημαντικό και το πιο ισχυρό εργαλείο στα πλαίσια τη εξωτερική πολιτική και πρέπει αυτά να τα βάλουμε μαζί. Δεν πρέπει απλώ να λέμε λίγα λόγια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουμε μια κανονική εμπορική σχέση με του Κινέζου. Όχι, πρέπει να ξανασκεφτούμε ε, θεμελιωδώ πώ αντιμετωπίζουμε την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Φρανσίσκο Χωσέ Μιλάν Ιμών για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε τρει πτυχέ εν συντομία ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση του COVID-19. Πρώτα απ' όλα, η κρίση αυτή απέδειξε, κατέδειξε τα προβλήματα που έχει σε υγειονομικό επίπεδο η διεθνή η παγκόσμια διαχείριση. Δεν μπόρεσαν οι αρμόδιε αρχέ να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ούτε την ανταλλαγή πληροφοριών, ούτε το συντονισμό ε, για την ε, ενημέρωση σχετικά με τον ιό. Επίση, υπάρχει τεράστια εξάρτηση τη Ευρωπαϊκή από το εξωτερικό. Χρειαζόμαστε ένα υψηλότερο επίπεδο υγειονομική αυτονομία. Δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα από τρίτε χώρε σε αυτό το βαθμό, σε στρατηγικού τομεί, όπω παραδείγματο χάρη το υγειονομικό υλικό ή ε, συστατικά ενεργέ ουσίε φαρμακευτικέ για την κατασκευή φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή 80% τη παγκόσμια παραγωγή αυτών των συστατικών ε, λαμβάνει χώρα στην Ινδία και στην Κίνα. Επίση είναι σαφές ότι πρέπει να βοηθήσουμε τι τρίτες χώρες, ιδιαίτερα τους, αφρικανικέ χώρε χώρες για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή. Και χαίρομαι που στην απάντηση της Ένωσης ε, υπάρχει μια σημαντική οικονομική συνεισφορά για την αντιμετώπιση τη πανδημία σε τρίτες χώρες. Και τέλος, ε, δυστυχώς, ε, ε, τις δύο τελευταίε ε, είχαμε δύο πανδημίες. Η δεύτερη πανδημία για κάποιο λόγο μας εξέπληξε. Είμαστε σε ένα παγκόσμιο ε, περιβάλλον και οι δεν ε, γνωρίζουν σύνορα. Την επόμενη οικονομική κρίση θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και πιο συντονισμένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χαβιέρ Λόπεθ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον είπα το εκπρόσωπο. Είναι αλήθεια ότι η πανδημία αυτή ε, δεν ήταν απλά η μεγαλύτερη πρόκληση του αιώνα ε, αλλά κατέδειξε και τις πολύ μεγάλες αντιφάσεις, τις μεγάλες αδυναμίες ε, ε, του μοντέλου παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ήταν αδυναμίες που τις βλέπαμε και πριν. Δεν υπάρχει ε, η ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολυμερείς, οργαν... Ε, πολυμερείς οργανισμοί είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένοι. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ένταση ε, στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Βεβαίως μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς πρέπει να δρούμε στο μέλλον. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει την ευθύνη ε, για να ε, υπάρξει μεταρρύθμιση των παγκόσμιων ε, ε οργανισμών. Για την κλιματική αλλαγή ε, για όλα αυτά χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Πρέπει να βρούμε και εμεί όμω το δικό μα ε, δρόμο για να υπερψηφιστούμε τι αξίε μα και τις, τα συμφέροντά μα στον κόσμο. Πρέπει να βρούμε συμμάχου ε, και να μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτού τι κρίσιμε στιγμέ. Η Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή ε, ζει την πανδημία αυτή με πολύ άσχημο τρόπο και πρέπει να είναι συμμαχό μα. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Γιορντάνοφ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, θα ήθελα να συγχαρούμε τους πολίτες του Χονγκ Κόνγκ, οι οποίοι ψώνουν τη φωνή τους για την ελευθερία τους μετά την απόφαση που πήρε το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας για τον νόμο εθνικής ασφάλειας. Εγώ εκπροσωπώ μια χώρα η οποία έχει εμπειρία από την φρίκη του ολοκληρωτισμού και γι' αυτό ζητάω από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλους τους ευρωβουλευτές να αποχαιρετήσουν τις ψευδεσίσεις μας ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι με την κομμουνιστική Κίνα. Πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτών του Χονγκ Κόνγκ. Οι αξίες μας απαιτούν από μας να πούμε στο καθεστώς του Πεκίνου ότι μπορούμε να σταματήσουμε την συμφωνία επενδύσεων και ότι είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε και μια πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Κίνας, όπως το κάναμε και μετά την ρωσική επίθεση κατά της Κρυμαίας. Οι κυρώσεις είναι και το μόνο μέσο το οποίο μπορεί να κάνει να λογικευτούν τέτοια κομμουνιστικά καθεστώτα τα οποία εξακολουθούν και ζουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η Μίριαμ Λέξμαν. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αν κάποιο δεν υψώσει τη φωνή του για την ελευθερία παντού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ελευθερία πουθενά. Η Κίνα ανατρέπει την αυτονομία του Χονγκ Κόνγκ, το κράτο δικαίου, τι θεμελιώδει ελευθερίε και τι διεθνεί συμφωνίε. Η τελευταία μονομερή απόφαση του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου τη Κίνα για ένα νόμο εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κόνγκ απειλεί σοβαρά την αυτονομία, το κράτο δικαίου και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Ο νόμος αυτός θα επιβάλλει διάφορα σαφή και δρακόντια μέτρα. Πριν από δύο εβδομάδες, 900 πολιτικοί ηγέτες μεταξύ αυτών και πολλοί από εσά, υπέγραψαν κοινή δήλωση καταδικάζοντα αυτή την ε, κίνηση. Και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασπάζεται τι αρχέ τη ελευθερία και βασίστε στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά το ΧΟΚΟΚ. Εμείς θα πρέπει την πολιτική μας να τη βασίσουμε στο άρθρο 21 της συνθήκης. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από όλες, όλους τους ευρωβουλευτές να στηρίξουν το ψήφισμα, όπως επίσης και τον λαό του Χονγκ Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ιζαμπέλ Σάντος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Από τότε που υπογράφτηκε η συνοβρετανική δήλωση όσον αφορά τη διακήρυξη όσον αφορά το Χοκόγκ, τότε αγνοούσαν πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως συνέβαινε σε ολόκληρη την Κίνα. Τώρα με τον νόμο αυτό για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι ότι αγνοεί το κράτος δικαίου και θέτει σε κίνδυνο την αρχή της μίας χώρας δύο συστήματα. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Η στρατηγική σχέση βέβαια ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι σημαντικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζητάμε λιγότερη συνοχή ανάμεσα σε αυτά που κάνουμε και τις αρχές μας. Αντίθετα, μας υποχρεώνει να απαιτήσουμε περισσότερο την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ και το διεθνές, την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Αυτά αναμένει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Χίλντε Φάτμαντς. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμε είπατε εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφέ ότι εγώ υποστηρίζω βεβαίω την αρχή μία χώρα, δύο συστήματα. Γι' αυτό και στηρίζω το λόγο του Χονγκ και την ελευθερία έκφρασή του. Είναι πολύ σημαντικό για οι δημοκρατικοί ηγέτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη του τι έγινε στις διαδηλώσει και τι σημαίνει για την αυτονομία του Χονγκ Κόνγκ αυτό ο νέο νόμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί και υπάρχει ένα πολύ έντονο ψηφισμό που ζητάει από την Κίνα να αποσύρει την νομοθεσία αυτή, να σεβαστεί την ελευθερία του λαού του Χονγκ Κονγκ και να δείξει ότι είναι έτοιμο να στηρίξει το κράτος δικαίου. Αλλιώς εμείς, η διεθνής κοινότητα, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως πάμε στο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μήπως εφαρμόσουμε κάποιο νόμο Μακνίσκι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι θα κάνουμε με τα κινέζικα προϊόντα. Νομίζω ότι μπορούμε με τόσα κινέζικα προϊόντα που εισάγουμε να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να επιμείνει για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Κίνα. Αυτό να το κάνουμε υποστηρίζοντα αρχέ και τι αξίε μα. Γι' αυτό κάνω και πάλι έκκληση Προ την Κίνα πρώτα απ' όλα. Να αποσύρει το νόμο για την εθνική ασφάλεια και να προσφέρει στο λαό του Χονγκ την αυτονομία η οποία έχει συμφωνηθεί με την συμφωνία μια χώρα δύο συστήματα. Σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει αξία και αρχές παντού στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στη Μάρα Μπιτζότο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κομμουνιστική Κίνα είναι πλέον η μεγαλύτερη απειλή στην ελευθερία και την δημοκρατία μας. Με τον κορονοϊό με την απειλή του Χονγκ Κόνγκ, με τους ε, Κινέζους κατασκόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, σκάνδαλο, είναι το ότι η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος και των Πεντεστέρων δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσει η σιωπή, τα παιχνίδια και τα ψέματα. Θα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια για τα εγκλήματα της Κίνας. Οι δικές μας αξίες δεν πολλούνται σε κάποιο βρώμικο εμπόριο αίματος. Λοιπόν, δεν πρόκειται μόνο για έναν οικονομικό πόλεμο, πρόκειται για έναν πόλεμο πολιτισμών τον οποίον κήρυξε κατά του δυτικού κόσμου η κινέζικη δικτατορία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε με όλα τα μέσα την ελευθερία και τη δημοκρατία μας. Οι Ιταλοί, οι Ευρωπαίοι, όλος ο κόσμος δεν θα γίνουν ποτέ σκλάβοι του κινέζικου κομμουνιστικού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει η Σίτα Κάνκο. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η επιτροπή αυτή υποσχέθηκε ότι θα είναι μια γεωπολιτική επιτροπή, όμως μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ανταυτού, βλέπω μια υπηρεσία εξωτερικής δράσης η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να κατευνάσει το Πεκίνο. Στην σύνοδο κορυφής επόμενης εβδομάδας είναι σαφές ότι οι Κινέζοι δεν θέλουν να σημειωθεί πρόβλημα